Τα αφορά για την κυκλοφορία οχημάτων εμπορευματικών μεταφορών. Τα πρωτόκολλα, τα, τα πρακτικά της 15ης ε, Δεκεμβρίου και της 16ης Ιανουαρίου και τα εγκεκριμένα κείμενα της 15ης Ιανουαρίου έχουν κοινοποιηθεί. Υπάρχουν ενστάσεις? Όχι, άρα θεωρείται ότι εγκρίνονται τα πρακτικά και τώρα περνάμε στο πρόγραμμα εργασίας. Όπως αποφασίστηκε στις 13 πρώτου ε, το πρόγραμμα εργασιών, η ημερήσια διάταξη ε, έχει διανεμηθεί και σας προτείνω να ε, παρατείνουμε τη σημερινή βραδινή συνεδρίαση μέχρι τις 9, όχι μέχρι τις 8 το βράδυ, μέχρι τις 9. Συμφωνείτε? Και τώρα προτείνω να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Προτού περάσουμε.